κυρία Άστον, σχετικά με το Κυργιστάν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Άστον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που έχω αυτή την δυνατότητα να κάνω τη δήλωση για το Κυργιστάν. Ε, όπως ε, γνωρίζετε όλοι εδώ οι περιστάμενοι, η κατάσταση παραμένει μάλλον ασαφής. Βεβαίως ε, το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και εγώ επανειλημμένα ασχολήθηκα με το θέμα. Επίσης, έστειλα αντιπροσωπέ υπό τον Πιέρ Μαρέλ επιτόπου έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένες επαφές επιτόπου. Η προσπάθεια που ε, ξεκίνησε στην πρωτεύουσα την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζεται ακόμη και βεβαίως η κρίση έχει ήδη δείξει τις επιπτώσεις της σε όλη την, ε, σε όλη την ε, περιοχή αυτή τη ε, στιγμή έλαβα και ένα μήνυμα ε, από τον απεσταλμένο, ο οποίος ε, μου λέει ότι τα πράγματα συνεχίζονται. Βεβαίως, η η αναχώρηση του Πρόεδρου από την χώρα οπωσδήποτε εκτόνωσε την κατάσταση και, θα την και η παρέτησή του και μετά η αναχώρησή του εκτόνωσε την κατάσταση και πιστεύω ότι θα την εκτονώσει περαιτέρω. Ε, χθες ε, μάθαμε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αναταραχές ε, και βεβαίως θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Θα πρέπει οι κάτοικοι του Κυργιζιστάν να συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή χωρίς μίσους αλλά και χωρίς φόβο για την ζωή τους. Όσον αφορά τώρα τον, το, την κυβέρνηση, την μεταβατική κυβέρνηση, ο κύριος Μπακίε βεβαίως έχει έχει παρατηθεί, αλλά θα πρέπει και η μεταβατική κυβέρνηση ε, να είναι νόμιμη. Αυτή τη στιγμή εκπονείται νέο σύνταγμα, το οποίο ε, θα αποτελέσει αντικείμενο δημοψηφίσματος και το Κοινοβούλιο ε, υπάρχει σχέδιο έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά όλη αυτή την δημοκρατική διαδικασία και όλα τα δημοψηφίσματα. Το σημαντικό είναι όλες οι παρατάξεις αλλά και όλες οι εθνοτικές ομάδες να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στα δημοψηφίσματα αυτά. Τα πρώτα δείγματα, κυρίε και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ενθαρρυντικά ε, και θα ζητηθούν ε, τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο σε επίπεδο Υπουργών. Βεβαίως, εάν ε, θέλει η χώρα να γυρίσει στην δημοκρατική, στη δημοκρατική οικογένεια, εμείς θα είμαστε ε, κοντά τους έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε. Ε, και φυσικά θα προσφέρουμε οποιαδήποτε τεχνογνωσία σε επίπεδο συντάγματος και νομοθεσίας με τον ΟΑΣΕ είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε έτσι ώστε να οργανωθούν σωστά οι επόμενες εκλογές. Ε, θα είμαστε κοντά στο Κυργιζιστάν έτσι ώστε ε, να ε, βρεθούν σωστές, ορθές, λογικές λύσεις για το μέλλον στο άμεσο μέλλον θα είμαστε στο πλευρό του Κυργιζιστάν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ε, προβλήματα ανθρωπιστικής φύσεως σε συνεργασία και με τον Ερυθρό Σταυρό. Φαίνεται πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μείζων ανθρωπιστικά προβλήματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μονάχα επιμέρους συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουμε την αρρωγή την οποία έχουμε ήδη ε, ξεκινήσει όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και την, ε, την καταπολέμηση της φτώχειας. 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στις ε, ταραχές του Μπίσκακ και πρέπει να πω ότι οτιδήποτε πρέπει να γίνει θα γίνει έτσι ώστε και τώρα και στο μέλλον να αποφευθούν τέτοιου είδες διαπραγματεύσεις. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ουσιώδης κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση γιατί εδώ έχουμε ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι κακές πολιτικές ε, επιλογές ε, μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτικά προβλήματα, ε, σε επιδείνωση της εγκληματικότητας, χαλάρωση των νόμων κλπ. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, θα είμαστε πάντα εδώ έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Και είμαι έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις σας για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Μπροκ. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την ε, εκτίμηση της κατάστασης και πράγματι πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκατασταθεί η τάξη, να διασφαλιστεί η ζωή των ανθρώπων και μετά τα υπόλοιπα, αλλά είναι σαφές ποια έκταση έχουν τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη που αποτελεί τη βάση της πολιτικής σταθερότητας. Και εδώ πέρα είναι ζήτημα ίσης μεταχείρισης που έχει καταστραφεί μέσω της διαφθοράς και αυτό απαιτέλεσε αιτία για την αντιπαράθεση αυτή. Επίσης πρέπει να δούμε πως οι χώρες αυτές είναι άσταθείς σε τέτοιο βαθμό ώστε οι προσπάθειές μας πρέπει να συνοδευτούν μέσω μιας οικοδόμησης του κράτους, δημοκρατίας και κράτους δικαίου και αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί ολόκληρη η περιοχή έχει στρατηγική σημασία όχι μόνο λόγω της ενέργειας, αλλά συνολικά. Εάν δούμε, παραδείγματο χάρη, τις ε, θρησκευτικές ε, πεπιθήσεις ε, των κρατών αυτών, οι οποίες στραφούν προς έναν φόντα θα έχουμε οδηγηθεί σε καταστροφικές συνέπειες. Οπότε η βοήθεια σε αυτές τις χώρες για να αποφευχθούν αυτές οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά σημαντική. Και για εμάς, για το δικό μας το συμφέρον, όχι μόνο για λόγους ανθρωπιστικούς. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι γείτονες έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για να μην εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή αδυναμίας για να ξαναξεκινήσουν τα παιχνίδια αυτά ισχύω που δεν ανήκουν στην εποχή μας. Για τρία λεπτά ο κύριος Βόμποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Απεσταλμένη, κυρία Υπερδιεκπρόσωπε. Ποια είναι η κατάσταση. Ένας δικτάτορας ή ένας δικτατορικός πρόεδρος πέφτει, η νεολαία χαίρεται για τη δημοκρατία και μετά από λίγους μήνες ξανά στα ίδια. Δηλαδή η δημοκρατία αποκαταστάθηκε για να έρθει ο γιος στην η κατάσταση καθώς από ό,τι φαίνεται Έχουμε ενδείξεις, αλλά οι ενδείξεις πλέον δεν αρκούν. Θέλουμε αποδείξεις. Εάν δεν θέλει ο τωρινός πρόεδρος να βρει την να έχει την μοίρα των προκατόχων του, πρέπει και ο ίδιος να αλλάξει στάση. Και από ό,τι φαίνεται πως δεν θα προσπαθήσει ξανά να δημιουργήσει διχόνοια αλλά θα προσπαθήσει να ζήσει στην εξορία και να αφήσει ήσυχους τους Κυργίζιους να οδεύσουν προς την δημοκρατία. Βεβαίως αυτά δεν ισχύουν μόνο στην Κυργισία αλλά και σε άλλες χώρες. Ευχόμαστε στον εκπρόσωπο του Καζακστάν καλή επιτυχία εξ του ΟΑΣΕ αλλά και στη χώρα του δεν είναι τόσο ιδιώδης η κατάσταση Ούτε στο Ουσμπεκιστάν επίσης τόσο ωραία τα πράγματα. Η δημοκρατία δεν είναι ένα πράγμα που το παίρνουμε και το κάνουμε εισαγωγή και το φέρνουμε κάπου. Οπότε πρέπει να παρακολουθήσουμε εδώ πέρα την όλη υπόθεση. Όπως είπε ο κύριος Μπρόκ, η όλη περιοχή είναι δύσκολη. Ο κύριος Μορέλ πράγματι ειδικό απεσταλμένος κάνει καλή δουλειά, αλλά δεν φτάνει αυτό, το θυμόμαστε ε, τι είχε γίνει και επί γερμανικής Προεδρίας είχε αναπτυχθεί επί, στα, επί κυρίου Στάινμαιρ μια στρατηγική για ολόκληρη την Κεντρική Ασία, την οποία θα πρέπει, δεν ξέρω, και εσείς να αναπτύξετε κάποιο, κάπως για να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή. Δεν είναι θέμα μόνο ενέργειας από το Τουρκμενιστάν μέχρι το Καζακστάν. Είναι θέμα σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στο Αφγανιστάν και σε κάποιες χώρες, Μπεκιστάν και λοιπές, ξέρουμε πως είναι επίσης ασταθής και προβληματική η κατάσταση. Είναι τελικά και θέμα ανθρωπιάς. Για τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία και με στοιχεία ανθρωπιάς και δημοκρατίας και να σπαρακαλώ παρακαλώ η Κυργυζία να αποτελέσει αφορμή Μία νέα στρατηγική εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβόμποντα. Ο κύριος Ρινάλντι για δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Αγαπητοί Συνάδελφοι, κυρία Ήπατη εκπρόσωπη, υπάρχει μια εξαιρετική ε, τελευταία ε, σελίδα στο τρομερό έπος του Κυργιζιστάν ε, που μας δίνει να καταλάβουμε και ποια είναι η ιστορία αυτής της χώρας όπου η σύζυγος του ήρωα που εκπροσωπεί ολόκληρο το έθνος προσπαθεί να προστατέψει τον τάφο του και αποφασίζει ότι δεν θα γραφτεί το όνομα του ήρωα μάνας ε, πάνω στον τάφο αυτό αλλά το όνομα της γυναίκας του έτσι ώστε να μην συλληθεί από τους βαρβάρους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε κι εμείς από τη νέα άρχουσα τάξη του Κυργιζιστάν που δεν είναι και τόσο νέα άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει εγώ λέω, βλέπω ότι υπάρχει επικοδομητική μάλλον θετική έστω και αν είναι ε, προσεκτική η στάση του Συμβουλίου και της, ε, είπα, της εκπροσώπου που όμως θα πρέπει να ζητηθούν συγκεκριμένα και σαφή ε, μέτρα μεταρρύθμισης. Όχι, όχι μόνο να υπάρχει σαφής οδικός χάρτης όσον αφορά την επανένταξη ε, δημοκρατικών ε, νόμων που θα έχουν επικυρωθεί και από την, τη λαϊκή φωνή αλλά οπωσδήποτε και μέτρα κατά της διαφθοράς έτσι ώστε να υπάρξει ανεξάρτητη ε, δικαιοσύνη που αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να καταργηθεί και αυτή η νομεκλατούρα η οποία είναι απολύτως γραφειοκρατική και η οποία στην ουσία ε, καταπιέζει τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το Κυργιζιστάν αντιμετωπίζει μια ε, κρίση και είναι μια καλή ευκαιρία ε, για να δοκιμάσουμε την ε, πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων στην Ασία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις χώρες αυτές να κυλήσουν σιγά σιγά στον ασφικτικό μάλλον εναγκαλισμό της Ρωσίας. Θα πρέπει να παίξουμε και εμείς τον ρόλο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούνατσα, για η κυρία Λούνατσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε και τι εκπρόσωπε. Ακούσαμε χτες πως είχαμε ελπίδες το 2005 με την Επανάσταση το νέο πρόεδρο που επιτέλους θα εκπροσωπούσε το λαό, θα είχαμε δημοκρατία, συμμετοχή. Βεβαίως όλα αυτά δεν προέκυψαν και συμβαίνει το ίδιο όπως κάνει το ίδιο ότι είχε κάνει και ο προκάτοχός του. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει μαζικά. Αυτό το απαιτούν οι καιροί και είπατε κυρία Άστον και χαιρετίζω το ότι ε, απεστήλατε αμέσως τον ειδικό εκπρόσωπο Μορέλ. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση από Δευτέρα ε, στο Συμβούλιο να ε, αναθεωρήσει τη στρατηγική της, ε, της Κεντρικής Ασίας για να είναι αποτελεσματική. Το ερώτημά μου είναι τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς θέλετε να υποστηρίξετε την διαδικασία του συντάγματος που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες όπως έχει προταθεί γιατί είναι αναγκαίο να συνεισφέρουμε στο ότι η περιοχή και η Κυργυζία να γίνουν ε, μια χώρα και ένας χώρος συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης. Ε, και αυτό είναι σημαντικό και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λουνάτσεκ. Ε, κυρία Βέρζια έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όντως η κατάσταση στην Κυριαζία είναι ασταθής. Ε, αυτή η χώρα ήταν μεταξύ αυτών που θεωρούσαμε πιο ανοιχτές για την δημιουργία δημοκρατικών θεσμών. Η επανάσταση των, του λοιπόν το 2005 δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες. Ο κύριος Μπασκεύ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πληθυσμού. Φαίνεται ότι πρόθεσε περαιτέρω την διαφθορά και συμμετείχε ο ίδιος ε, αλλά και η οικογένειά του αδειάζοντας τα ταμεία και δημιουργώντας μάλλον επιβάλλοντας ένα σύστημα πολύ πιο καταπιστικό. Μετά από τις ε, εξέγεση της ε, 17 Απριλίου ε, μια προσωρινή κυβέρνηση ανέλαβε τα ενία, αλλά ο κ. Μπάσκεφ φαίνεται ότι δεν παρετήθηκε ακόμα και αν εγκατέλειψε την ε, χώρα. Νέε εξεγέρσει έλαβαν χώρα χθε, όπω το είπατε, στο νότο τη χώρα και γύρω-γύρω από την πρωτεύουσα. Κύριε Επίτροπε, αυτή η χώρα έχει σημαντική στρατηγική σημασία και όχι μόνο σε, ε, στο επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι το πεδίο αντιπαράθεσης ε, μερικών μεγάλων δυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα καλά λόγια, δεν είναι ιδιαίτερα παρούσα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Η υποστήριξή της, η διευρωπαϊκή της παρουσία είναι χαλαρή. Αρκεί να διαβάσουμε τα... την ενημέρωση η οποία φτάνει από... Ε, ώρα με την ώρα βλέπουμε τις σχέσεις που έχει το Καζακστάν και με τη Ρωσία. Αλλά η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της χώρας. Έχετε δίκιο, κυρία είπατε εκπρόσωπος. Θα πρέπει να αποκατασταθεί το κράτος αλλά πολύ γρήγορα θα πρέπει να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε μια πραγματική στρατηγική για αυτή την περιοχή του κόσμου. Ναι, Πρέπει να βοηθήσουμε την χώρα να καταπολεμήσει την ένδυα. 40% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, χρειάζεται να διευκολύνουμε την οικονομική ανάπτυξη και όπως το δηλώσατε, ιδιαίτερα σε ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας, αλλά και σε ζητήματα νερού, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τις περιοχές. Πρέπει να υποστηρίξουμε φυσικά τη δημοκρατία και την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα αυτό είναι απόλυτα κατεπήγον. Ε, η δέσμευσή μας θα πρέπει να είναι να εμποδίσουμε τη χώρα αυτή να κατρακυλήσει προς τον ολοκληρωτισμό και ένα νέο αυτορχικό καθεστώς. Δεν ε, αρκεί να ε, αναμειχθούμε στα εσωτερικέ υποθέσει του, εναντίον να βοηθήσουμε του Κυργίζιου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Αυτό είναι το κλειδί προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ε, έναν ρόλο κινητήριο σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ, κυρία ο κύριος Προβέρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο, στην Κυριαζία είναι πολύ σημαντική για την σταθερότητα στην Κεντρική Ασία με περιοχή στην οποία η Ευρώπη έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα οποία αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και ενέργεια. Μετά από την αρχέ τη 7 η Απριλίου χρειάζεται να αποκαταστήσουμε στις συνθηκε προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε ένα δημοκρατικό καθεστώ μέσω ελεύθερων ε, εκλογών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μας ενισχύει το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό όπλων έχει διαφύγει μέσω λαθρεμπόρων και συμμοριών και να, μπορεί να τροφοδοτήσει την τρομοκρατία στην περιοχή και τις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει παράλληλα με, την, με τον ΟΑΣΕ ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε σταθερές και δημοκρατικές ε, αρχές ε, και διαδικασίες. Δεν μπορούμε να έχουμε την ψευδέστηση ότι ένα νέο σύνταγμα ή ένα κοινοβουλευτικό καθεστώ θα οδηγήσει απαραίτητα στη δημοκρατία. Θα πρέπει να οριμάσουν οι πολίτες και να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτό τον τομέα και για ένα μεγάλο διάστημα εμεί θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Προδέρα. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Βαϊντέρου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα οι ταραχές οδήγησαν την Κυργιζία σε μια πολιτική, οικονομική και οικονομική κρίση. Διαδλήθηκε ουσιαστικά το συνταγματικό δικαστήριο, εμφανίστηκαν διάφορες ε, προσωρινές κυβερνήσεις, ενώ ο πρόεδρος Μπακίεφ λέει πως πλαστογραφήθηκε η υπογραφή του και δεν έχει παρετηθεί. Εν τω μεταξύ προσπαθούν διάφορες κυβερνήσεις να αναλάβουν περιφερειακές διοικήσεις και εθνικές ε, συσπυρώσεις δημιουργούν φόβο εθνοτικής βίας. Ε, συμμορίες ε, λειτουργούν ελεύθερα, κυκλοφορούν όπλα και γίνονται ληστείες. Η ασφάλεια και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών εκεί πέρα κινδυνεύουν. Οπότε δεν μπορεί η ενδιάμεση κυβέρνηση να αντιμετωπίσει καμία από αυτές τις απειλές και δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους ντόπιου. Η κυρία Άστον εξέδωσε δηλώσεις εκφράζοντας την ανησυχία της αλλά χρειάζονται πράξεις και πιο ενεργά βήματα. Πρέπει να λάβει αποφασιστική στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση στη χώρα στην πάρα πολύ σημαντική αυτή η χώρα. Πρέπει να είμαστε πιο παρόντες, συνεργαζόμενοι με τον ΟΗΕ, της ΗΠΑ και τον ΟΑΣΕ για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υπερασπίσουν τη ζωή και την περιουσία τους. Είναι σαφές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει μια ανεξάρτητη έρευνα για τις αιτίε και τα αποτελέσματα των ταραχών Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί η, τράπεζα, η Κυργιζιανή Τράπεζα Ανάπτυξης ε, και βοήθεια πριν δοθεί οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Επίσης δεν υπάρχει πραγματική στρατηγική κατά το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες εξελίξεις και να υποβαθμίσει τα ίδια τα συμφέροντα και την αξιοπιστία της Ένωσης στην περιοχή και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την συνάδελφο για δύο λεπτά. Το λόγο έχει η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέδι Αστόν, στα 20 χρόνια της ανεξαρτησίας του το Κυργιστάν κυβερνήθηκε από διεφθαρμένα καθεστώτα και ελάχιστη πρόοδο έγινε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δημοκρατικών θεσμών. Όσον αφορά τα τελευταία 15 χρόνια, μπορώ να σα διαβεβαιώσω έχοντας και προσωπική εμπλοκή ω εκ τη ιδιότητας μου του ΑΣΕ και άλλο πώ. Οι άνθρωποι που κυβερνούσαν μέχρι χτέ, και οι άνθρωποι που του ανέτρεψαν είναι όλοι του συστατικά του ιδίου διεφθαρμένου συστήματο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο στρατό βρίσκεται μέσα στην Πισκέκ, την πρωτεύουσα, και κάνει έρευνε και συλλήψει. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην παρούσα διακυβέρνηση, διότι είμαστε στο, τελευταίο στάδιο πριν από τον εφήλιο και πριν από τον διαμελισμό τη χώρα ο λαό του Κυργιστάν είναι ένα φιλιρινικός λαό και φαντάζομαι αρκετοί από εσά θα τον έχετε γνωρίσει μέσα από τα βιβλία του διάσημου συγγραφέα του Τζιγκί Αϊτμάτοφ που ήταν πρέσβη στι Βρυξέλλε μέχρι και πριν από τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η οικονομική δυσπραγία και οι κοινωνικέ ανισότητε, καθώ επίση και οι παρεμβάσει ξένων χωρών προκαλούν εκρήξει που μπορούν να φτάσουν καμιά φορά στα όρια του εμφυλίου πολέμου και εδώ θα διαφωνήσω λίγο αν ο λαό του Κυργιστάν μπορεί να εκτρέψει την τρομοκρατία όπως είπα ο κίνδυνος διαμελισμού του κυργιστάν σε βόρειο και νότιο είναι υπαρκτός και καλλιεργείται από ξένους παράγοντες ενώ η συμμετοχή της χώρας στον οασε και η συνεχής παρουσία του οασε στο κυργιστάν δεν φαίνεται να έδωσε καρπούς προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. βεβαίως υπάρχει μια μόνιμη ανθρωπιστική κρίση μπορεί να μην είναι οξία η ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει αλλά ε, δεν έχει επέλθει κανένας εξυγχρονισμός και καμία βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών όλα αυτά τα χρόνια και ο κόσμος ζει πολύ πιο κάτω από τα όρια τη φτώχεια. γι' αυτό είναι απαραίτητο να παρέμβει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σε συνεννόηση με του λοιπού θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιτροπή και το συμβούλιο και να αναθεωρηθεί η στρατηγική που ακολουθείται μέχρι σήμερα στην περιοχή. Ε, μια ισχυρή αντιπροσωπεία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου πρέπει να παρακολουθήσει την πορεία εκδημοκρατισμού και να χορηγεί τα κονδύλια με ελεγχόμενο τρόπο με στόχο την ανάπτυξη των θεσμών και τη παιδείας γιατί η αποσταθεροποίηση του κυργιστάν συνιστά μείζωνα κίνδυνο για αποσταθεροποίηση σε όλο τον χώρο τη Κεντρική και τη πρόσω Ασία αλλά και τη Ευρώπη. εάν δε η ευρωπαϊκή ένωση θέλει να διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό ειρηνευτικό ρόλο πρέπει να δράσει τώρα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και θα δώσουμε το λόγο αμέσως στην κυρία Μπασέσκου η κατάσταση στο Κυργιστάν είναι εξαιρετικά ανησυχητική λόγω της γεννητική θέσεως που κατέχει στην Ασία. Πρόκειται για αμερικανική βάση με πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Επίσης ε, σταθμεύουν εκεί και ε, ρωσικές ε, δυνάμεις, στρατιωτικέ δυνάμεις. Την προηγούμενη εβδομάδα χάθηκαν ανθρώπινε ζωέ λόγω των αναταραχών και θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τις ε, τελευταίες ημέρες ε, υπήρξαν ε, νέες αναταραχές ανάμεσα σε Κυργισίους με Κυργισιανή κατάσταση καταγωγή ε, Τούρκους και Ρώσους. Οι εθνοτικές διαμάχες συνεχίζουν ε, και μπορεί να αποσταθεροποιηθεί ολόκληρη η περιοχή. Πρέπει επομένως να προσέξουμε ιδιαιτέρως ε, αυτήν την κατάσταση στο Κυργιστάν και να βοηθήσουμε τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιμπο Μπάιντελ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Άστον. Σήμερα μιλάμε για τα ανησυχητικά συμβάντα στο Κυργιστάνα και ε, προσπαθούμε να βρούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ε, φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή και να κάνουμε την κατάσταση πιο σταθερή. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά την εξομάλυνση της ε, κατάστασης ε, και έτσι ώστε να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ε, ζωές. πρέπει να προστατέψουμε τη ζωή των κατοίκων των πολιτών του Κυργιστάν. Βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις, να υπεραμεινθούμε και των δικαιωμάτων των φυλακισμένων πολιτών Σαράουι. Κοιτάξτε, όσοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο θα μιλήσουν, λέει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό λίγη υπομονή μονάχο. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ανησυχητικά τα πρόσφατα γεγονότα στο Μπισκέπ και είναι θλιβερό τέλος για την επανάσταση της του Λίπας και αντί βεβαίως για δημοκρατία τι μας έδωσε ο πρόεδρος νεποτισμό και αυταρχισμό υπάρχει εδώ πέρα στην κοιλάδα Φεργάνα διείσδυση ε, ακραίων Ισλαμιστών τα τελευταία χρόνια και βέβαια υπάρχει και η κυβέρνηση ο Τονπάγεβα, η οποία από ό,τι φαίνεται στρέφεται προς την Ρωσία η οποία υποστήριξε την ανατροπή του προηγούμενου καθεστώτος. Η δε κυρία Τομπάγεβα είχε υπηρετήσει ως πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε ξέρει τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η περιοχή είναι σημαντική για λόγους και ασφάλειας και ενέργειας. Γνωρίζουμε και την αεροπορική βάση των ΙΠΑ, η οποία υποστηρίζει την δύναμη που βρίσκεται στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πέντε χρόνια μετά την επανάσταση της, ε, των, του λοιπόν η κατάσταση έγινε πραγματικά ιδιαίτερα προβληματική. Εντάξει, γιατί, αυτό, διότι υπάρχει νεποντισμό, δεν υπάρχει δημοκρατικό κράτος, υπάρχουν οικονομικές φύσει, προβλήματα και άλλα. Θεωρώ πως ε, η πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε ότι δηλαδή ο κύριος Μορέλ θα έχει την δυνατότητα να μας ενημερώνει για την κατάσταση στο ε, Κυργυζία είναι μια πρωτοβουλία που θα πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερα συμφέροντα. Θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου η χώρα αυτή να παραμείνει δημοκρατική. Πάνω από 80 θύματα υπήρξαν. Αυτό είναι ένα πολύ κακό μήνυμα. Χρειάζεται η αποστολή του απεσταλμένου μας να ε, στεφθεί υπό Το λόγο έχει ο κ. Πρέγα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Κυργιστάν δεν είναι δυστυχώς ο έσχατος των ηγετών που απογοητεύει τους πολίτες του. Αυτό το οποίο <clears throat> βλέπουμε είναι ότι χωρίς σταθερούς και υγιείς δημοκρατικούς θεσμούς καμία χώρα δεν μπορεί να προοδεύσει ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ρωσική στρατιωτική βάση και μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Κυργιζία και συχνά χρησιμοποιούσαν ως όπλο τον εκβιασμό για να πετυχαίνουν περισσότερα προνόμια από τους μεν και τους δε. Αλλά τώρα χρειάζεται να σταματήσουμε τη βία. Η βία θα πρέπει να λήξει το συντομό των δυνατών. Διότι ενώ υπάρχει βία δεν μπορεί να υπάρξει ένα νέο σύνταγμα. Το λόγο έχει ο κύριος Τσίμπετ. Σιλβέστερς. Η κατάσταση στο Κυργιστάν είναι οπωσδήποτε επικίνδυνη, τουλάχιστον ε, και σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, γιατί φαίνεται ότι ε, πηγαίνει όλο και περισσότερο προς την τελωνιακή και οικονομική επιρροή της Ρωσίας η χώρα αυτή. Ξέρουμε ότι άλλαξαν τα πράγματα τον, στα, στις 15 Απριλίου όταν έφυγε δηλαδή ο, πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός αλλά ε, δεν ξέρουμε προς τα πού ε, και ακόμα όμως δεν έχει παρετηθεί και ακριβώς απαιτώντας την παρέτησή του κατέβηκαν οι άνθρωποι στον δρόμο. Πρόκειται για μια χώρα ε, η οποία ναι, μεν είναι μικρή, αλλά ε, το μόνο ε, λειτουργών νοσοκομείο που έχει είναι σε μια ξένη στερεωτική βάση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε πάση θυσία να αποφευχθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Όλα αυτά κυρία Άστον τα αναφέρατε εσείς και είπατε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε. Ναι, να βοηθήσουμε σε δύο μέτωπα και στο διπλωματικό με μέτωπα, αλλά όπως και εσείς η ίδια είπατε κυρία μου, ε, σε συγκεκριμένο απτό και υλικό επίπεδο, δηλαδή να δώσουμε βοήθεια ε, η οποία θα μειώσει, αν όχι αφανίσει, οποιοδήποτε στοιχείο κοινωνικής αναταραχής. Εδώ δεν είμαστε στην ΑΕΤ, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είμαστε στο Κυργιστάν, να σπάσουμε τουλάχιστον στην ώρα μας. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο και την επόμενη φορά σα παρακαλούμε να μιλήσετε λίγο πιο αργά, ε, γιατί διαφορετικά θα έχουν μεγάλα προβλήματα οι διερμηνείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση νόμιζαν κάποιοι πως η δημοκρατία θα έρθει από μόνη της. Σήμερα γνωρίζουμε πως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος που βαρύνει αυτές τις χώρες από την εποχή των Σοβιέτη, των Σοβιέτ. Καθώς επίσης και πράγματα τα οποία είχαν καταπιεστεί πολιτισμικές και σκεφτικές φορές οι οποίες έρχονται στο φως και όλα αυτά θα κοστίσουν στην χώρα αυτή και σε άλλες. Από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με φήμες υπήρξαν ξένοι μισθοφόροι οι οποίοι πυροβόλησαν τον κόσμο στους δρόμους του Μπισκέκ. Από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να διεθνοποιήσουν την ε, σύγκρουση και βεβαίως αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία της περιοχής και για την ατοική και τη γερμανική αποστολή στο Αφγανιστάν. Οπότε θα πρέπει εδώ πέρα πρώτα απ' όλα και για τη δημοκρατία να καταπολεμήσουμε και την διαφθορά και τις τοπικές φατρίες. Μόνο τότε υπάρχει κάποια ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Μπέναράτ. Μπέναράτ. Ε, Κυρία, ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό σχέδιο ανοίγει μια νέα και φιλόδοξη αρχή. Αυτή η ε, ψηφιακή βιβλιοθήκη θα μας βοηθήσει στο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας η συμμετοχή των χωρών σε αυτό το σχέδιο είναι σημαντική. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν αφορά και μια θεμελιώδη αρχή αυτή της πολιτιστικής διαφοράς και στόχος μας είναι ε, η Αφρικανική Ήπειρος. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, έχουμε μάλλον την υποχρέωση να αναγνωρίσουμε την συστήση ε, αυτού του, αυτών των λαών. Μπορούμε, χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να καταστήσουμε τους ε, Αφρικανούς ε, ικανούς ε, να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση της, του πολιτισμού τους στην Αφρική. Λέγεται ότι κάθε ηλικιωμένος που αποθνίσκει είναι μια βιβλιοθήκη που χάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία με ανθρωπολόγους της Αφρικής κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στο να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την ε, πολιτιστική ποικιλότητα της ε, Ιφιλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο για τα συμπεράσματα στην κυρία Άστον που είναι η πατή εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ο τίτλος της στην οθόνη διότι εκτός από το είπατε εκπρόσωπος είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να μπει ο πλήρης τίτλος λοιπόν. Ορισμένοι βουλευτές έκαναν πάρα πολύ σωστές και ορθές παρατηρήσεις. Ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Τάνοκ και λοιποί μίλησαν για την φτώχεια της χώρας αυτής, μία από τις φτωχότερες της ε, Κεντρικής ε, Ασίας. Και βεβαίως εμείς σαν Ευρωπαίοι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές. Ε, συμβάλλουμε περισσότερο δηλαδή στο κατακεφαλήν εισόδημα και οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε κι άλλα έτσι ώστε να εκριζωθεί η φτώχεια. Ο κύριος Σβόποντα είπε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει στη χώρα αυτή μια ουσιαστική πολιτική αναμόρφωση σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ ε, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αυτές τις μέρες βρίσκεται επί τόπου επ' αυτού εργάζεται και βεβαίω για να προσπαθήσει να αποτρέψει οποιαδήποτε συνέχεια ή επανάληψη των ταραχών. Βεβαίω υπάρχει μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική αυτή μέσα στα πλαίσια ε, της στρατηγικής ε, της ομάδας εξωτερικής δράσης και να δούμε τι μπορεί να κάνει και το Συμβούλιο. Ο κύριος Μανάλτη και άλλοι ε, είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε θετικοί, επικοδομητικοί και προσεκτικοί ταυτοχρόνως. Συμφωνώ και θα συμφωνήσω και με όλους όσους αναφέρονται στην σημασία της επιβολής του νόμου να υπάρξει ε, σωστή εφαρμογή του νόμου, να υπάρχει σωστό νομικό ε, σύστημα και βεβαίως να προωθηθεί και η αναμενόμενη και τόσο απαραίτητη μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία σειρά πραγμάτων. Βεβαίως ε, οικονομική βοήθεια, ε, στήριξη στην ε, νομική και συνταγματική και πολιτική μεταρρύθμιση, εφαρμογή του νόμου ε, βεβαίως αυτό που αναφέρατε για τη διαχείριση των υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες είναι πλούσιες σε υδάτινους πόρους και επομένως ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία την οποία κάναμε και πριν από πέντε χρόνια όσον αφορά την βοήθεια ε, σχετικά με τη διαχείριση των ε, δημάτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο Πιέρ Μοράλε ήταν επιτόπου αρκετές μέρες και μόλις ε, γύρισε. Στις 27 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα εμφανιστεί η ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να ε, μιλήσει και για την ε, αποστολή του εκεί. Και φυσικά έρχεται σε και επαφή με όλους τους συναδέλφους του. Είμαστε λοιπόν παρόντες, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, ξεπεράσουμε ε, ε, να ξεπεράσουμε οποιασδήποτε φήμες για αστάθεια, οποιασδήποτε φήμες και να, να μείνουμε στα πραγματικά γεγονότα. Ελπίζω ότι ε, σύντομα θα είμαστε σε θέση να πάρουμε και πιο συγκεκριμένα βήματα. Κοιτάξτε, ορισμένα από τα παρόντα μέλη του κυβερνητικού σχηματισμού ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στην αντιπολίτευση ε, και ε, το αυταρχικό καθεστώς του ε, Προέδρου τους είχε πραγματικά υποδιωγμό. Αυτό από μόνο του υπόσχεται πολλά για την περιοχή. Βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους πολιτικούς αυτούς έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες συνταγματικές και νομοθετικές αλλαγές οι οποίες θα προετοιμάσουν ένα σωστό μέλλον. Θα συνεχίσουμε και τη στρατηγική μας έτσι όπως την ε, έχουμε εκπονήσει μέχρι τώρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Άστον, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής ε, και τη εκπρόσωπε. Ακούσαμε με προσοχή τα όσα μας είπατε για την Κυργυζία. Τώρα θα, ακούσουμε, θα σας ακούσουμε την ίδια προσοχή να μας μιλάτε για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Ε, να σας πω ότι Έχω δεχθεί τρεις προτάσεις ψηφίσματος ή μάλλον